ψηφίσματος για το Κονγκό. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Ψηφοφορία για έξι προτάσεις ψηφίσματος για το ΛΕΠΑΛ. Έχουμε κάποιες προφορικές τροπολογίες από τον κύριο Ρωμέ Βερουέδα. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Έχω αρκετέ προφορικέ τροπολογίε. μπορώ να τις διαβάσω όλες μαζί και μετά να τις ψηφίσουμε unblock. Ε, η A και η C, αντικατάσταση Civil War με την ένοπλη σύραξη. Δεύτερον, να βάλουμε αντί για PLA Former Maoist Combatants. Στο D, το terminate by abolish the monarchy να αντικατασταθεί και πάλι abolish the monarchy στο 8, στο 9 να αντικαταστήσουμε το CPN κάθετος N με το UCPN κάθετος N στο K να αντικαταστήσουμε το other με το close to και να προσθέσουμε και το 30% και να προσθέσουμε και το one off στην παράγραφο 1 να λέμε at the permanent constitution, στο 15 να αφαιρέσουμε το τελευταίο τμήμα της φράσης regrets however that its status as an independent body has not been uh, ratified by law και τέλος να διαγράψουμε τον όρο revolutionary στο 18. Αυτές είναι όλες οι προφορικές τροπολογίες. Έχω την αίσθηση ότι συμφωνούν όλοι με τις τροπολογίες, απλώς ε, θα ήθελα να καταγραφούν τα πρακτικά. λογικά υπάρχουν στον κατάλογο. Δεν είναι στον κατάλογο, μου λένε, αλλά λογικά πρέπει να τις έχετε τις προφορικές τροπολογίες. Λογικά έχουν διανεμηθεί σε ομάδες, οπότε τις έχουν όλοι. Υπάρχουν ενστάσεις για τις τροπολογίες αυτές. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν τις προφορικές τροπολογίες. Θα τις ψηφίσουμε αμπλεκ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Παράγραφος 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε τώρα το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τέλος, έχουμε έξι προτάσεις ψηφίσματος για τη Λιβύη. Ονομαστική κλίση για το σύνολο του ψηφίσματος. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Και ο κύριος Πόσελτ ακόμα. Μάλιστα. So, Ε, τότε ψηφίσαμε όλοι, άμα ψήφισε και ο κύριος Πόσελτ. Πέρασε. Εγκρίνεται. Now I still have some statements to make. Έχω ακόμα μερικές δηλώσεις να σας κάνω. Τα χαρτιά μου είναι στα τσεχικά και θα τα διαβάσω τσεχικά. Θα ήθελα να σας πω ότι η κυρία Ζανίν Χένης Πλάσχαρτ και ο κύριος Πακέ μας διαβίβασαν γραπτός ότι ε, ε, παρετούνται από